Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που είστε τόσο πολύ άριθμοι σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Μια συνεδρίαση που δυστυχώς έχει βαριά σκιά από το τραγικό δυστύχημα των μαλαισιανών αερογραμμών στην Ουκρανία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και συνεδρίες των συντονιστών, αλλά θέλω πρώτα ξεκινώντα να απευθύνω ένα φόρο τιμής και συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να γερθούμε όλοι σε ένδειξη σεβασμού για ένα λεπτό. Wir kommen dann zu unserer Tagesordnung. Θα περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Την έχετε λάβει και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Αλλιώς συγκρίνεται. Έχετε επίσης τα πρακτικά στη διάθεσή σας. Και πάλι αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνονται. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντίρρηση. Τώρα, αποφάσεις των συντονιστών. Από εδώ και μπρος θα γίνονται γραπτός, θα καταγράφονται γραπτός τα συμπεράσματα της, των συντονιστών. Θα τα λαμβάνετε εγκαίρως σε γραπτή μορφή και θα, μπορείτε, θα μπορούμε να τα συζητούμε. Τώρα λοιπόν θα τα συζητήσουμε μέχρι τις 3 το απόγευμα, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, μέχρι τις 3 η ώρα όπως είπα, μπορούμε να πούμε ότι ε, εγκρίνεται από το Ινολβέρια της Επιτροπής και το κείμενο των συντονιστών. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Καλώς. τα έγγραφα. Καταρχάς έχουμε το πακέτο καλωσορίσματος της Επιτροπής μας, πολλά καινούργια μέλη όπως ξέρετε, και για αυτούς τους συναδέλφους, τους νέους συναδέλφους έχουμε ετοιμάσει ένα φάκελο με τα απαραίτητα για το κολοσόρισες έγγραφα με αυτό υπενθυμίζουμε και στους νέους συναδέλφους αλλά και στους παλιούς, αν χρειάζεται, τι έχουμε κάνει τελευταία πενταετία. 2009-2004 λοιπόν, 2014 έχετε την ε, επισκόπηση των κύριων νομοθετικών μας έργων. Και η Γενική Διεύθυνση MOVE, ε, μεταφορών δηλαδή, με τον Επίτροπο Κάλλας, θα είναι σήμερα το απόγευμα μαζί μας για να μας παρουσιάσει ε, και το μελλοντικό πρόγραμμα και τον απολογισμό. Και θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε στην πενταετή στρατηγική της ε, υπηρεσίας ΕΜΖΑ για τις θαλάσσιες μεταφορές, ένα έγγραφο το οποίο έχει κατατεθεί Μα καλεί σε επίσκεψη η ΕΜΖΑ. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε σε μεταγενέστερη συνεδρίαση. Αυτά λοιπόν τώρα για τι πρώτε διατυπώσει και τώρα θα περάσω στο πρώτο σημείο της της διάταξης και θα καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά τον Υπουργό Μεταφορών της Ιταλικής Προεδρίας, τον κύριο Λούπη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπουμε εδώ. Κύριε Λούπη, έχετε το λόγο για να μας εκθέσετε τις, προεδρίες, τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Grazie signor Presidente. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους ευρωβουλευτές που είναι παρόντες σε αυτή την ε, επιτροπή και με ιδιαίτερη χαρά αλλά και μεγάλη αίσθηση ευθύνης θα σας παρουσιάσω σήμερα στην Επιτροπή της Προτεραιότητας της Ιταλικής Προεδρίας στον τομέα των μεταφορών. Η Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, συμπίπτει με μια στιγμή πολύ σημαντική για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι πολλές οι άγνωστες συνιστώσεις, αλλά είναι και πάρα πολλές οι ευθύνες ε, που έχουμε όλοι μας έτσι ώστε το μέλλον να καταστεί όλο ένα και πιο βέβαιο και πιο σίγουρο. Καταρχήν, η πρώτο άγνωστος ε, χ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη, σε κάθε μια χώρα, είναι η ελπίδα της ε, μιας στεναρής και στέρεης ανάκαμψης μετά από τόσα χρόνια παραταμένης κρίσης η οποία έχει διαδώσει, έχει τροφοδοτήσει μια μεγάλη αίσθηση αντιευρωπαϊσμού που φάνηκε και στις τελευταίες ευρωεκλογέ. Για να μπορέσουμε, πρέπει να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. θα πρέπει από κοινού με την επόμενη Κομισιόν να υιοθετήσουμε μια ημερήσια διάταξη που να ε, προωθήσει την ανάπτυξη, τη βιώσιμη, τη σταθερότητα και τη συνοχή. Παράλληλα θα πρέπει να ανανεωθούν ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι σχέσεις τους με τα κρατη Και σε αυτή την προοπτική θα πρέπει να δούμε την Ιταλική Προεδρία. Ένα κίνητρο και φιλοδοξίες, φιλόδοξη στόχη μέσω του συντονισμού με τα κρατημέλη. Ανάπτυξη και απασχόληση είναι ε, δύο ανάμεσα στις ε, κύριες προτεραιότητες του Ιταλικού Εξαμήνου της Προεδρίας. Ανάπτυξη και απασχόληση είναι στόχοι αλλά και η δέσμευση που η Κομισιόν από κοινού με το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβουν και μόνο μέσω μιας συγκεκριμένης μαρτυρίας για το πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη και για την απασχόληση, για την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας στην Ευρώπη θα μπορέσουμε πραγματικά να αποδείξουμε την εγκυρότητα και την ισχύ του μεγάλου ευρωπαϊκού ονείρου. Ο τομέας των υποδομών και των μεταφορών είναι θεμελιώδης σε την οπτική. Το θέμα που θέλουμε και πρέπει να θέσουμε ως Προεδρία Ιταλική αυτού το εξάμεινο είναι το πώς οι μεταφορές και οι υποδομές θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία, μια μεγάλη όθηση για να ανακάμψει η ανάπτυξη αλλά και η απασχόληση αλλά και η αξιοπιστή ολόκληρης της Ευρώπης και η πραγματική ένωση στην Ευρώπη. Δεν γίνεται ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτό. Διακόπτει ο υπουργό. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Εντάξει, δεν έχουμε μόνο στην Ιταλία τεχνικά προβλήματα. Α proposito τη Όσον αφορά τις υποδομές λοιπόν, έλεγα ότι το δίκτυο μεταφορών της Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει την ανταγωνιστικότητα και τη συνογή και να σέβεται υψηλά στάνταρ βιωσιμότητας και ασφάλειας. Οι πολιτικές μεταφορών θα πρέπει να είναι συνεπείς με τους στόχους της απομάκρυσης του άνθρακα από την ευρωπαϊκή οικονομία. Πολύ συχνά ε, βλέπουμε τραγικά γεγονότα τα οποία ε, πλήττουν τους Ευρωπαίους πολίτες στη διάρκεια των μεταφορών, της μετακίνησής τους. Η ασφάλεια θα πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο από την πρόβλεψη, το σχεδιασμό των δικτύων μέχρι τη λειτουργικότητα των ε, μέσων μεταφορών. Υλικά και άλλα προσόντα που θα έχουν τα μέσα μεταφοράς ε, στις ε, αστικές αλλά και στις υπαίθριες μεταφορές ε, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν δεν γίνουν οι επενδύσεις που προβλέπονται θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ρήξη με το παρελθόν. Καταρχήν θα πρέπει να ξεπεράσουμε το παράδοξο της δημόσιας οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της περίοδου 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στην αξιοσημείωτη δέσμευση της Επιτροπής Επιτροπής και στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο ε, είχα, θα καλύψει περίπου 27,4 από τα 250 δις που προβλέπονται ως επενδύσεις για την υλοποίηση ε, των ε, προγραμμάτων TNT και των ψηφιακών υποδομών. Το υπόλοιπο κόστος σε μεγάλο βαθμό θα επιβαρύνει τους προπολογισμού των κρατών μελών που παρόλα αυτά εμποδίζονται λόγω των λοιπών πόρων και λόγω των δεσμεύσεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε αυτό το σημαντικό θέμα οι υποδομές για την ανάπτυξη θα αφιερώσει η, Ευρωπαϊκή, Ιταλική Προεδρία το, το άτυπο συμβούλιο που θα γίνει ανάμεσα στους Υπουργούς ε, Μεταφορών και στο Μιλάνο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Σκοπεύουμε να προωθήσουμε τον ορισμό μιας κοινή θέσης για τη μεγαλύτερη ευελιξία από πλευρά των κρατών μελών, των ε, δημοσίων συνεισφορών αλλά και των διευθυντικών ταμείων για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα σημαντικά διευρωπαϊκά, μάλλον διασυνοριακά ε, δίκτυα. Σκοπεύουμε επίση να αντιμετωπίσουμε και το θέμα τη διακυβέρνηση των διαδρόμων για να καταστεί πιο αποτελεσματική διαχείριση. Όσον αφορά του πόρου, του ιδιωτικού είναι σημαντικό να κάνουμε έναν απολογισμό των όσων πετύχαμε την περασμένη δεκαετία και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε χρηματοδότηση από την αγορά. Τα μέσα, τα καινοτόμα όπω ε, το Ταμείο Μαργαρίτα και άλλα μέσα δεν έχουν βρει ακόμα, δεν ε, τα ομόλογα έργου δεν έχουν βρει ακόμα την κατάλληλη του εφαρμογή. Τόσο λόγω ε, αμοιβή, ε, όσο και λόγω προβλημάτων ρυθμιστικών. Τέλος, ακόμα και η εφαρμογή της Ευρωβινιέτ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Έχουμε δηλαδή εδώ 15 με 25% αύξηση συγκεκριμένων οδικών ε, τμήματων υπέρ διαφόρων ε, ε, τρόπων μεταφοράς ε, ε, έχουν εφαρμοστεί τελικά μόνο στην Αυστρία. Η ρήξη λοιπόν με το παρελθόν αφορά και τη διακυβέρνηση των προγραμμάτων τέντια Μέσα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου για κάθε διάδρομο θα υιοθετηθεί ένα σχέδιο εργασίας με περιγραφή συγκεκριμένων μέτρων για κάθε χώρα ώστε να αρθούν τα γεωγραφικά, τεχνικά, λειτουργικά και διοικητικά εμπόδια και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μεταφορών και των πολυτροπικών μεταφορών. Έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το περιεχόμενο των μεμονωμένων σχεδίων εργασίας κατά τη διάρκεια του ατύπου Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου, θα προωθήσει η Ιταλική Προεδρία μια σύγκριση ανάμεσα στα διάφορα μέσα διακυβέρνησης των διαδρόμων. Αυτά όλα ευνοούν την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να ισχύσουν και ορισμένοι όροι. Ο πρώτος συνδέεται με την ακύρωση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στις ισχυρές και στις αδύναμες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική θα πρέπει να φροντίσει για την συνοχή με την ίδια ισχύ, όπως και ασχολείται και με την οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε επίσης ε, διάφορα μποτιλιαρίσματα, τα οποία προκαλούνται από συγκεκριμένα προβλήματα στις, ε, σε συγκεκριμένες περιοχές και μπορεί να εμποδίσουν τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έπειτα θα πρέπει να δούμε την ε, μείωση του κόστους ε, το, το, το, της υλικοτεχνικής υποδομής όσον αφορά την αξία της παραγωγής, το κόστος της μεταφοράς όσον αφορά τα μεταφερόμενα αγαθά ε, αντιστοιχεί στο 12% και μπορεί να μειωθεί στο 8% μόνο εάν βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή. Αυτό σημαίνει ανάκτηση πάνω από 180 δις ευρώ. Αυτό αποδεικνύει πως χρειάζεται ε, νέα στρατηγική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα δίκτυα μεταφορών. Αυτοί οι όροι μας επιβάλλουν να επεξεργαστούμε έναν κώδικα δεοντολογίας που θα πρέπει να χαρακτηρίσει ολόκληρο το εξάμεινο αλλά και τη νέα θητεία ολόκληρη. Θα πρέπει να είναι ένας κώδικας που θα περιλαμβάνει κάνει διάφορους στόχους. Ο πρώτος είναι η εναρμόνιση των χρονικών διαστημάτων όπου τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν ε, αυτή την ε, οργανωτική και ουσιαστική, το ουσιαστικό σχέδιο για τις υποδομές. Θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή ένα συγκεκριμένο οικονομικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο. Έχουμε ε, χρηματοδοτήσει τις δομές CORE, τα δίκτυα TEN, αλλά θα πρέπει να συντονιστούν οι χρόνοι αλλά και οι τρόποι εφαρμογής όλων αυτών των προγραμμάτων. Δεν είναι μόνο ο προγραμματισμός η πρόκληση, αλλά και η υλοποίηση όλων αυτών των προτεραιοτήτων που έχουμε θεσπίσει. Το δεύτερο κριτήριο στόχος θα πρέπει να είναι ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους πόρους ενώπιον των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μα, η συμβολή των μεμονωμένων χωρών, ε, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία. Όπως Πώς θα γίνει όμως ε, στην εφαρμογή η συμβολή αυτή, πώς ε, θα επηρεάσει τους πόρους που στόχο έχουν την επίτευξη του στόχου, δηλαδή την υλοποίηση των 10T. Η δεύτερη σχετίζεται με τη σχέση των πόρων σε μια συγκεκριμένη λογική κοινή ωφέλεια, δηλαδή ανάγκη να δημιουργηθεί ένα, κυλιό, ένα κυλιόμενο ταμείο όσον αφορά τι ε, κοινοτικέ χρηκοδοτήσει. Τέλος, ε, έχουμε να κάνουμε με την ε, συμμετοχή των ιδιωτικών κονδυλίων. Αυτό θα ενισχυθεί μόνο εάν οι ιδιώτες πιστούν πως θα έχουν απόδοση. Μόνο με τέτοιο τρόπο θα μπορέσουν να πάρουν σάρκα και οστά τα ομόλογα έργο. Το Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου θα είναι και μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε την ε, αστική κινητικότητα. Είναι μια από τις κύριες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλική Προεδρία αποδίδει σε αυτό το θέμα και διόλου τυχαία το έχει εντάξει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών που θα γίνει στο Μιλάνο. Θεωρεί λοιπόν πως είναι ένα σημαντικό θέμα. Τη στιγμή που υλοποιούνται τα μεγάλα δίκτυα σύνδεσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρειάζεται οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που που εστιάζονται στους αστικούς κόμβους και στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές των χωρών μας. Η ε, ε, αστική ενότητα είναι η πρόκληση του μέλλοντος. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε συνδυάζοντας νέες τεχνολογίες, την δυνατότητα νέων μέσων που επιτρέπουν να σεβαστούμε το περιβάλλον αλλά και να διευκολύνουμε τη σύνδεση και τη μετακίνηση με πιο ταχύ τρόπο. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, για να αυξηθεί η ε, απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα χρειάζονται διευθυντικά ταμεία τα οποία θα στηρίξουν κάθε τρόπο μεταφορά. Ε, η Ιταλική Προεδρία θα συζητήσει και θα εγκρίνει συγκεκριμένα νομοθετικά ντοσιέ που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Τέταρτο πακέτο για του σιδηροδρόμου. Αντιπροσωπεύει σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνοντα την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περασμένη θητεία συνέβαλε σημαντικά σε όλα αυτά έτσι ώστε να φτάσουμε στον ορισμό και ε, του τετάρτου σιδηρονομικού πακέτου. Το Συμβούλιο Υπουργών αλλά και η Κομισιόν αντιμετώπισαν και όρισαν τα στοιχεία τα οποία αφορούν το τεχνικό πυλώνα αυτού του τετάρτου σιδηροδρομικού πακέτου. Παραμένει ακόμα ανοιχτό το θέμα της διακυβέρνησης και του ε, πολιτικού πυλώνα, τη διακυβέρνηση, το άνοιγμα της αγοράς αλλά και συγκεκριμένη πτυχή που εγώ θεωρώ ότι πρέπει πολύ προσεκτικά να το εξετάσουμε ως κρατημέλη και αφορά λοιπόν την πτυχή ε, της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αλλά και της περιφερειακής. Η Ιταλία δεσμεύεται από αυτή την άποψη λοιπόν να εργαστεί σε συνεργασία με όλα τα κρατημέλη ώστε να επιταχύνει τις εργασίες και την πρόοδο αυτών Προχωρώντας στον ορισμό των τριών φακέλων που περιλαμβάνουν και αποτελούν, συναποτελούν τον τεχνικό πυλώνα που ορίστηκε από το Συμβούλιο των Μεταφορών υπό την Ελληνική Προεδρία και να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Επιπλέον, επειδή το τέταρτο συνδρομικό πακέτο είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν και τα θέματα του πολιτικού πυλώνα, χρειάζεται και επιθυμούμε να αρχίσουμε να συζητάμε τα κράτη-μέλη και με το Κοινοβούλιο και όλο ένα και περισσότερο ε, το περιεχόμενο αυτής της διακυβέρνησης και του πολιτικού πυλώνα. Στον ε, πολιτικό πυλώνα θεωρούμε πως η διαφάνεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ε, σωστή διακυβέρνηση πριν ακόμα από τον διαχωρισμό ε, της ιδιοκτησίας. Για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους το κράτος οφείλει να αναφερθεί στα πρότυπα holding λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταρρυθμίσεις σε κάποια καρδιμαλή. Επίσης θεωρούμε πως η ισορροπία και η παρακολούθηση των σχέσεων ανάμεσα στους διαχειριστές των υποδομών και της υδροδομικής εταιρεία από τη στιγμή που έχει υπάρξει λογιστική αλλά και επιχειρησιακή διάκριση θα είναι αυτό το θέμα ρύθμισης εξάντε ε, όσον αλλά και εξ Η επαλήθευση των ε, θεμάτων ανταγωνισμού έχει στόχο να μην υπάρξουν διακρίσεις, να υπάρχει ποιότητα στις υπηρεσίες, ε, τιμές να είναι προσιτές και να υπάρχουν παροχή του αγαθού και της υπηρεσίας υπό διαφανείς συνθήκες. Όσον αφορά την υποχρέωση ε, υπηρεσίας κοινωνικής οπέλης, δημόσιας υπηρεσίας, θα πρέπει να ενεργήσουμε με ομοιογενή και βέβαιο τρόπο με συγκεκριμένα προκαθορισμένα πλαίσια. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένο ανταγωνισμό, θεμητό ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο όσον αφορά τις υπηρεσίες της αγοράς, αλλά και τις δημόσιες τοπικές ε, αγορές ε, που έχουν γίνει εμπορικές υπηρεσίες μόνο σε κάποια κράτη-μέλη, ενώ κάποια άλλα κράτη-μέλη έχουν μείνει πίσω και έχουν καθορίσει ανομιγενές πλαίσιο τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εμποδίζει συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνισμού. Θα χρειαστεί λοιπόν ως προς αυτό να σκεφτούμε ποιο είναι, θα είναι το εύρος μιας τέτοιας απελευθέρωσης, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τη λεπτότητα και την ευαισθησία καθώς και το βασικό ρόλο που παίζουν οι τοπικέ δημόσιε υπηρεσίε σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Ιταλία που ήδη έχει εμπειρία απελευθέρωσης όπως και άλλα κρατημέλη θεωρεί πως η αμοιβαιότητα είναι ο βασικός δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να καταστεί δυνατό ένα σύστημα αυτορύθμισης της αγοράς. Εξάλλου, όσον αφορά τις δαπάνε τη δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να ξεπεραστεί ο, ο κατακαιρματισμός του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, όσον αφορά δε τη μεταφορά των επιβατών ε, ε, για των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα πρέπει να καταστεί διαφανής και η διαδικασία ε, προκήρυξης διαχωνισμών, ώστε το κοινό να μπορέσει να προσαρμοστεί όμω Θα πρέπει να υπάρξουν και κατάλληλε προθεσμίε. Σκοπεύουμε λοιπόν να κάνουμε τη σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα του πολιτικού και τη διακυβέρνηση. Είμαστε πεπισμένοι ότι συνεπής και συνεκτική ανάπτυξη καθώς ε, μια ενιαία αγοράς του σιδηροδρομικού τομέα θα πρέπει να βασιστεί στα μοντέλα holding που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τον ενιαίο ε, ευρωπαϊκό ουρανό, βρισκόμαστε σε καθοριστική φάση. Το περασμένο Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια νομοθετική πρόταση που στόχο έχει να τροποποιήσει και να ε, προωθήσει τους τους, τις ρυθμίσεις όσον αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτό το νομοθετικό πακέτο το πακέτο ε, ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 2 θα έχει σημαντική επίπτωση όσον αφορά ολόκληρη την βιομηχανία θα αντιμετωπιστούν κρίσιμα σημεία τα οποία έχουν αναγνωριστεί από όλου του ενδιαφερόμενου φορεί και που αυτή τη στιγμή περιορίζουν τα ωφέλη του ενιαίου ευρωπαϊκού, που απορρέουν από έναν ενιαίο ευρωπαϊκό αγορό. Θέλουμε να έχουμε ε, ανταγωνιστική αεροπορία και να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που προκύπτουν από την αυξημένη ε, κυκλοφορία, ενέργεια κυκλοφορία που προβλέπεται για τα επόμενα έτη. Η Ιταλική Προεδρία θα ε, προτείνει μια επικοδομητική προσέγγιση που θα αξιοποιεί τις θέσεις που έχουμε μέχρι στιγμής και θα βοηθά στο να επιτευχθούν οι στόχοι του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δε συνέβαλε σημαντικά επειδή ενέκρινε τον περασμένο Μάρτιο μια σημαντική τροποποίηση των κυμάτων που επιλύουν κάποια από τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει τα κράτη-μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Η, Ευρωπαϊκή, η Ιταλική, με συγχωρείτε, Προεδρία έχει εντάξει τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό μόνο δύο ανάμεσα στα θέματα προτεραιότητας του εξαμήνου της Προεδρίας, ακριβώς επειδή θέλει να αντιμετωπίσει θέματα κλειδιά, διευκολύνοντας μια συζήτηση για συγκεκριμένα θέματα και να δώσει έτσι μια περαιτέρω όθηση στην υλοποίηση του συστήματος ΣΕΖΕΡ και στην επίτευξη των στόχων του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Με, στόχο, με αυτό το στόχο έχουμε προβλέψει μια έκθεση προόδου το Συμβούλιο της 8 η Οκτωβρίου που θα ακολουθήσει στις 6 και 7 Νοεμβρίου με υπουργική, ε, υπουργική ε, ε, σύνοδο για το θέμα αυτό που θα διοργανωθεί μαζί με την Κομισιόν στη Ρώμη. Στοχό είναι να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το τομέα και ευχόμαστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα γενικό προσανατολισμό στο Συμβούλιο τη 3 η Δεκεμβρίου ε, που με βάση τα αποτελέσματα τη Ρώμης. Τώρα όσον αφορά τι οδικές μεταφορέ, είναι στόχο τη Προεδρία να προχωρήσουμε από το Σεπτέμβριο στην εξέταση τη πρώτη οδηγίας για το Cross-Border Enforcement στην έδρα τη ομάδα εργασία του Συμβουλίου καθώ και θα ξεκινήσουμε τι επαφέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες να φτάσουμε σε τριμερή διάλογο και σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά το βάρος και τις μάξιμουμ διαστάσεις των εμπορικών οχημάτων που κυκλοφορούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία σκοπεύει να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υιοθέτησε στις 15 Απριλίου 2014 τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση για να επαληθεύσει τις δυνατότητες ε, επίτευξη συμφωνία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα στη διάρκεια ενό τριμερού διαλόγου. Αυτό θα επέτρεπε να υιοθετηθεί η οδηγία σύμφωνα με την επιταχυμένη διαδικασία έγκρισης στη δεύτερη ανάγνωση. Για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι πολύ σημαντική η ρύθμιση όσον αφορά τις ε, λιμενικές υπηρεσίες. Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο πιο συγκεκριμένα έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ασχολούνται μάλλον με το θέμα αυτό. Η αναθεώρηση των δικτύων TNT δημιούργησε τη βάση για μια νέα κατεύθυνση στην λιμενική πολιτική και έχει εντοπίσει τις μελλοντικέ γραμμές ανάπτυξης όσον αφορά ολόκληρο το δίκτυο μεταφορών της Ευρωπαϊκή Ένωση με μια πολύ επιλεκτική στρατηγική. Αυτή στην όπω όπως και στην Ευρώπη, είναι πια η στιγμή της επιλογής. Επιλογών που πρέπει να γίνουν αξιοποιώντας τους βασικούς στρατηγικούς κόμβους και δίνοντας ε, έμφαση στην υλικοτεχνική υποδομή ώστε να υπάρξει επαρότητος συντονισμό για να μπορούν τα εμπορεύματα να ταξιδεύουν μέσα από αποτελεσματικούς διαδρόμους και με μεγαλύτερη ταχύτητα, όσο γίνεται μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα λιμάνια και οι η σύνδεσή τους είναι πολύ σημαντικά ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών μεταφορών ε, και να τις συντονίσουμε καλύτερα. Και ακριβώς γι' αυτό η Κομισιόν έχει ορίσει τα λιμάνια ως ε, κινητήρες της ανάπτυξης. Η Ιταλική Προεδρία σκοπεύει να προωθήσει την πρόταση Κομισιόν με στόχο να οριστούν κοινές, ε, κοινοί και να αποφευχθούν ε, να αποφευθεί μάλλον αθέμητος ανταγωνισμός και να ε, ε, χρειάζονται περισσότεροι μάλλον κανόνες ε, πιο συνεπείς για να αναρμονιστούν οι νομοθεσίες που ισχύουν με σεβασμό όμως στις εθνικές ιδιαιτερότητες. Είμαστε πεπισμένοι πως πρέπει να εντοπιστεί ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο αναφοράς, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει χωρίς να θυσιαστούν οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Ευχόμαστε να υπάρξει αποτέλεσμα, ε, ικανοποιητικό αποτέλεσμα για όλα τα κατημέλη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το συμφέρον ενό τομέα το, αυτό το τον, λιμενικό που μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο για την Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, αξιότιμοι συνάδελφοι, η φιλοδοξία μας είναι να συμβάλλουμε μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και την ε, ασφάλεια ε, και μάλλον και την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορές να ενισχύσουμε την αγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση στην Ευρώπη των ανθρώπων, των οικογενειών, των ε, επιχειρήσεων. Περισσότερο από ποτέ οι πολίτες ζητούν αποτελέσματα και επιλογές που θα δώσουν, θα μαρτυρήσουν ότι περισσότερο καλύτερη Ευρώπη σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, το να επιδιώξουμε αυτό το στόχο είναι ηθικό μας καθήκον αλλά και πολιτικό. Σας ευχαριστώ. Herr Minister Lupi, vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir sind jetzt Σας ευχαριστούμε θερμά για την εισήγηση, κύριε Υπουργέ. Είμαστε ενήμεροι λοιπόν τώρα για, το σχέδιο, για τα σχέδια της ε, Ιταλικής Προεδρίας. Θα ακολουθήσουμε τη σειρά με τους συντονιστές πρώτους από τρία λεπτά, τις ομάδες από δύο, τους συναδέλφους δηλαδή από δύο, ανάλογα με τις ομάδες και μετά θα ξαναδώσουμε το λόγο στον ε, Υπουργό. Παρακαλώ, κύριος Φαντενκάμπ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και καλημέρα σε όλους. Κύριε Λούπη, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με μεγάλη χαρά περιμένει τη συνεργασία με την Ιταλική Προεδρία, έστω και αν σε ορισμένα ζητήματα μπορεί να υπάρξουν πιο δύσκολες καταστάσεις. Προς το παρόν, οφείλω σήμερα να αναφερθώ στην τραγωδία που έλαβε χώρα την προηγούμενη Πέμπτη στην Ουκρανία και να ρωτήσω εάν το Συμβούλιο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ασχοληθεί με την κατάρριψη του αεροσκάφους ή τι είδους πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αναλάβει το Συμβούλιο. Ξέρω ότι ίσως είναι κάπως νωρίς. Αλλά έχουμε τόσα θύματα και εκεί τους θρυνούν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπάρξει κάποια αντίδραση. Και για να περάσω τώρα στο πρόγραμμα της Τελικής Προεδρίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα χρειαστεί ασφαλώς πολλές αντοχές για να υλοποιηθεί. Αλλά όπως λέμε στην Ολλανδία, οι καλές προθέσεις μόνο δεν αρκούν. Χρειάζονται και ε, απτά αποτελέσματα. Ερωτώ λοιπόν τον Υπουργό ως πρόσωπο της Προεδρίας τι διδάγματα αποκομίζει στην πρώτη αυτή επαφή που είχε με το αντικείμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέλαβε τη σκητάλη από την ελληνική προεδρία, έχει ένα εξάμεινο, μας λέει ότι θέλει μέσα στο εξάμεινο να υλοποιήσει το τέταρτο πακέτο για του σιδηροδρόμους. Πολύ ωραία. Πώ όμω θα το υλοποιήσετε αυτό, Πώ, Ή μπορείτε να πείτε από κάποια μηνύματα που ενδεχομένω έχετε λάβει ότι θα τα καταφέρετε μέχρι τα Χριστούγεννα φέτος να το κλείσετε. Έχετε δει κάποιες ε, τοποθετήσεις από κυβερνήσεις Φερρυπίν. Λοιπόν, τις καλές προθέσεις τις βλέπουμε και τις αντιλαμβανόμαστε και τις βάζουμε και στα εγγραφά σα. Αλλά θα θέλαμε πιο συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Για τα θέματα των ε, αερολιμένων τώρα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς, θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να μας, να μας αναφέρετε, να μας εκθέσετε το χρονοδιάγραμμα που έχετε προβλέψει για να αντιμετωπίσετε το ακαθόδες αυτό ζήτημα. Και τρίτο ακαθόδες ζήτημα βέβαια οι λιμενικές υπηρεσίες και η διαφάνεια, η οικονομική διαφάνεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στους λιμένες δεν έχω καμιά ε, επιφύλαξη ως προς τη γνησιότητα των προθέσεων και των, των προσπαθειών σας, αλλά συγκεκριμένα τι πρόοδο περιμένετε να υλοποιήσετε μέσα στους έξι επόμενους μήνες και σύντομα μερικά σχόλια, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά αυτά που ακούσαμε για τους σπόρους, για τους διαδρόμους TNT, αλλά ας είμαστε και προσεκτικοί ως προς την ευελιξία. Σε περιόδους κρίσεως μπορεί η ευελιξία να φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική ιδέα, αλλά μπορεί τελικά να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες δαπάνες, ενώ εμείς το ΕΛΚ θέλουμε να περικόπτουμε τις δαπάνες για τους ε, οδηγούς. Πολλά ακούγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ οδηγών από διαφορετικές χώρες. Δεν ξέρω αν η Ιταλία έχει το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίσει, αλλά θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Κράμερ. Ο κύριος Ερτού έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σας χαιρετίζω εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι και προσδοκώ πολύ καλή συνεργασία. Μπορείτε να στηρίζεστε σε εμά και σας διαβεβαιούμε για την υποστήριξη που σας προσφέρουμε. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων. Ιδιαίτερος χαιρετίζω τις προσπάθειες της Προεδρίας σας για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει και για τη συνέχιση εκείνων που χρειάζεται να συνεχιστούν σε όλους τους τομείς των μεταφορών. Ιδιαίτερα αναφερθήκατε εσείς στον χώρο των σιδηροδρομικό. Έχουμε, όπως ξέρετε, να αντιμετωπίσουμε εδώ και τεχνικά ακόμη προβλήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υπόθεση αυτή και να εξασφαλίσουμε μια ενιαία αγορά. Αυτά λοιπόν τα τεχνικά ζητήματα. τα προωθείτε και δεδομένου ότι θεωρώ ότι στα τεχνικά ζητήματα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να βρούμε μια λύση παρά μεταξύ πολιτικών, το ξέρουμε αυτό άλλωστε στην Ευρώπη είναι πολύ πιο συνηθισμένο, θα ήθελα λοιπόν ε, να ξαναδούμε το θέμα αυτό το φθινόπωρο στην Επιτροπή μας και γι' αυτό θα ήθελα να ε, δω τι είδους προσδοκίες έχετε για επιτυχία σε τεχνικά αυτά ζητήματα η οδηγία 9653 που έχει να κάνει για τις, με τις μετρήσεις για τα φορτηγά οχήματα έχει να καταγράψει μια σειρά από τεχνικά επιτεύγματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν όμως ε, τεχνικά επιτεύγματα και πρόοδος ως προς τις προδιαγραφές τεχνικές, φερρυπίν, αεροδυναμικά στο όχημα, προδιαγραφές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ε, με την, κατανάλωση, με την καλύτερη κατανάλωση καύσιμου. καυσίμου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δω πώς εσείς δεσμεύεστε και πώς μπορεί το Συμβούλιο στο σύνολό του να ακολουθήσει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα ώστε να προχωρήσει το νέο ε, κείμενο αυτής της οδηγίας ώστε να ε, αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα όπως η παραδείγματι η πολύ μακρά κατεμέ μεταβατική περίοδος της οκταετίας που προβλέπεται σε αυτήν. Ένα άλλο ζήτημα που έχει ε, καταστεί πλέον μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πεπαλαιωμένες, ταλαιπωρημένες υποδομές των μεταφορών, γέφυρες και το καθεξής. Ερωτώ λοιπόν εάν έχετε κάποιες συγκεκριμένες προθέσεις και ποιες είναι αυτές, εάν μπορούμε να περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από την Ιταλική Προεδρία στους προσεχείς μήνες. Και για να κλείσω, χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφερθήκατε στα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα. Έχουμε και εμείς πολύ μεγάλη σημασία αποδόσεις σε αυτά και πρέπει να υλοποιηθούν πλέον ε, οι αποφάσεις και τα μέτρα. Κατά τα άλλα στη διατύπωση ίσως ε, κάποιο πρόβλημα ε, ως προς την διατύπωση να υπάρχει, γιατί εμείς δεν είχαμε ζητήσει αλλαγή ορισμού, δηλαδή δεν ζητούμε να αλλάξει η, η, η επιβάρυνση των οδικών μεταφορών σχέση με τις σιδηροδρομικές. Το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τσίλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών. Εγώ εκπροσωπώ την ομάδα μεταρρυθμιστών και συντηρητικών και προσβλέπω σε πολύ επικοδομητική και καρποφόρα συνεργασία. Ε, ο κύριος Βαντενκάμπ μας ανέφερε το θέμα ε, το, της συντριβής του αεροσκάφους και πιστεύω ότι στα θέματα αυτά το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών θα πρέπει να αποφανθεί κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιήσουμε μερικές ε, διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη και την συντριβή του αεροσκάφους που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς είναι δυνατόν ε, αρχηγός ενός κράτους ε, να λέει ότι όλη την ευθύνη τη φέρει η χώρα στην οποία έλαβε χώρα αυτό το ατύχημα. Μπορεί νομικά να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορεί μια χώρα να, ελέγχει. Η συγκεκριμένη χώρα δεν έλεγχε την, την τοποθεσία στην οποία έλαβε χώρα αυτό το ατύχημα. Θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη από το Συμβούλιο Μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Το σιδηροδρομικό πακέτο. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και αντιλαμβάνομαι ότι σας ενδιαφέρει η διεκπαιρέωση του θέματος αυτού στο Συμβούλιο προκειμένου να βρεθεί μια νέα προσέγγιση ομοιόμορφη και να καλύπτει η προσέγγιση αυτή και τις κοινοφέλης υπηρεσίες και αν ε, δεν συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι το τέλη Οκτωβρίου τουλάχιστον να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο για τα τεχνικά ζητήματα. Ερμήνευσα σωστά τις προθέσεις για το σιδηροδρομικό πακέτο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ενέργειες μεταφορές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται ε, στα θέματα αυτά και εξετάζει με μεγάλη σοβαρότητα τα θέματα. Ελπίζω να σημειωθεί κάποια πρόοδο και από το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση Connecting Europe και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, πιστεύω ότι και στον προπολογισμό μας θα πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα και τα σχέδια που καλύπτονται από το Connecting Europe Facility, αυτή τη διευκόλυνση του συνδέοντα στην Ευρώπη, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Γιατί άλλο ήταν το μήνυμα που ακούσαμε μέχρι στιγμή από τον προπολογισμό. Γιατί φαίνεται ότι περικόπτονται πολλά προγράμματα από, από τη διευκόλυνση αυτή. Κάτι τέτοιο θα έδινε ένα αντιφατικό μήνυμα και θα υπονόμευε μακρόπνοα σχέδια μεταφορών. Επίσης, θα ήθελα να μας διευκρινίσετε αυτά που είπατε στην ορισμό που δώσατε για την Ευρωπαϊκά Δικτύα Μεταφορών. Ε, ενιαία δίκτυα ε, οδικών, σιδηροδρομικών μεταφορών και λιμενικών. Θα τροποποιήσετε τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο έγγραφο και που αποτέλεσε τον καρπό μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων. Σας εύχομαι πάντως καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή τύχη και επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζήλα. Η κυρία Μάισνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό, τον κύριο Λούπη, που ήρθε για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας. Είμαι μπροστά σας κύριε Υπουργέ και εκπροσωπώ τους φιλελεύθερους. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο τρίλεπτο που δικαιούμαι. Κύριε Υπουργέ, μας μιλήσατε για τις προτεραιότητές σας, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Αυτά είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που μας απασχόλησαν και στο παρελθόν. Και, μια, και έχουμε και το Connecting Europe Facility, αυτή τη διευκόλυνση του στην Ευρώπη, πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Μιλήσατε για κάποιες προθεσμίες εκτέλεσης. Πολύ ωραία. Αλλά έχουμε και την αρχή use it or lose it. Δηλαδή ή το χρησιμοποιείς ή χάνεις την ευκαιρία αυτή. Επίσης έχουμε τα project bonds, τα ομόλογα έργα, ε, μια πολύ καινοτόμα μορφή χρηματοδότησης. Τα αναφέρατε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ομόλογα έργου και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια πιο ενισχυμένη συγχρηματοδότηση για να βρούμε περισσότερα κονδύλια. Το θέμα του ορισμού, το σχολείο ο κύριος Έρτοκ. Είναι νομοθετικό το θέμα και σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό πακέτο είπατε ότι θέλετε να ε, διεκπαιρεώσετε το πακέτο ενιαίο, ως ενιαίο πακέτο πολύ ωραία και αξιέπαινη προσπάθεια, αλλά αν δεν ευοδοθεί τουλάχιστον να διευθετήσουμε τα τεχνικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά του ενιαίου ευρωπαϊκού εθέρε, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, μιλήσατε για μια επικοδομητική πρόταση. Θα μπορούσατε να μα δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε. Γιατί αυτά που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμή δεν έχουν εφαρμοστεί. Κάτι που δεν είναι πρωτοφανέ. Με ενδιαφέρει όμω το πώ θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Εγώ είμαι Γερμανίδα και μερικές φορές γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα διασύνδεσης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, ενώ ε, η διασύνδεση Γαλλίας-Ιταλίας ε, λειτουργεί καλύτερα. Έχετε κάποιο σχόλιο σχετικά. Σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές, μας είπατε ότι θα πρέπει διασυνοριακά να εφαρμοστεί η ενωσιακή νομοθεσία. Μιλήσατε για τις διαστάσεις και το βάρος των οχημάτων, πολύ ωραίο. Παραλείψατε όμως μερικά σημεία που κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, μια ολοκληρωμένη ε, πολιτική για τη θάλασσα, κάτι που προϋποθέτει και τις θαλάσσιες μεταφορές. Μιλήσαμε για τη γαλάζια ανάπτυξη. Για παράδειγμα, παράκτιος τουρισμός. Γιατί και ο τουρισμός είναι ένα θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Δεν ξέρω αν είναι και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, αλλά το θέμα της ε, ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, για το ναυάγιο του Κώστα Κονκόρδια. Έχετε να μας πείτε κάτι, γιατί αυτές τις μέρες έγινε η ανέλκυση του ναυαγίου. Επίσης, τι γίνεται με τους επιβάτες ε, στις αεροπορικές μεταφορές. Νομίζω ότι τήρησα το τρίλεπτο που είχα στην διάθεσή μου. Έτσι δεν είναι. Σχεδόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ο Ματέο Ρέντζι, ο Ιταλός Πρωθυπουργός, είπε στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ένας από τους στόχους της Ιταλικής Προεδρίας, εδώ είμαι κύριε Υπουργέ, είναι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη μετά από λίγους μήνες θα γίνει ε, στο Παρίσι το 2015 η Διεθνής ε, Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να συμμετέχει και το μέσο των μεταφορών στην προσπάθεια καταπολέμησης της θέρμανσης του πλανήτη. Επίσης ε, θα ληφθούν υπόψη ενέργειες μεταφορές προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίμα. Μιλήσατε για αβιώσιμε μεταφορέ, μεταφορές, μεταφορέ. μεταφορές. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ποιο είναι όμως το φιλοπορία σας σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την ε, χρηματοδότηση μεγάλων μακρόπρων προγραμμάτων που κατά τη γνώμη μου είναι άχρηστα. Και θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λιόν Τουράν, το, η σύραγγα αυτή, Τουρίνο Λιόν. Έχουμε πολλές και διάφορες μελέτες για, για το έργο αυτό. Για το, τη σύραγγα αυτή Λιόν Τουρίνο, ποιε είναι οι προβλέψει χρηματοδότηση, ε, ποιε είναι οι προβλέψει κόστου, και πώ θα το λάβει αυτό υπόψη, ποιε είναι οι στάσει τη τελική προεδρία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Και όταν μιλούμε για μακρόπνοα αλλά άχρηστα σχέδια, θα ήθελα να ρωτήσω πώ ε, σκοπεύετε να καταπολεμήσετε τη διαφθορά, ιδιαίτερα στα μείζωνα σχέδια υποδομών και τι προσπάθειες θα γίνουν για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η δωροδοκία. Και δύο ακόμη ερωτησούλες προς τον Υπουργό πριν εξαντλήσω το τριλεπτό μου. Μας είπατε ότι οι μεταφορές αγγίζουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ιταλική Προεδρία τι σκοπεύει να κάνει προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις μεταφορές που θα πρέπει να είναι και ποιοτικές να ε, εξασφαλίζεται διατροπικότητα και να είναι και ποιοτικέ οι μεταφορές, να υπάρχουν συχνές ε, συνδέσεις. Επίσης, ε, τι γίνεται με το ποδήλατο, με τις αστικές συγκοινωνίες. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς τους δύο κλάδους ώστε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες που υπάρχουν στις μεταφορές και να ελαφρύνουμε κάπως τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Επίσης, πώς θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα, κυρίως η αποτελεσματικότητα των υποδομών, που άλλες φορές παρουσιάζουν ελλείψεις και άλλες φορές ε, πλεόνασμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κάρι Μαντελή. Και τώρα, τελευταίο συντονιστή, ο κύριο Λούμικρεν. Ευχαριστώ πολύ. 30 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα των μεταφορών και κυρίως των σιδηροδρομικών. Βλέπουμε λοιπόν στις μεταφορές ότι στη Σουηδία έχουν επιδεινωθεί σημαντικά οι συνθήκες, ιδιαίτερα στις οδικές μεταφορές, με την εισαγωγή της ε, ελεύθερης αγοράς ε, επιδεινώνονται οι συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα γίνεται λόγος για πράσινες μεταφορές, αλλά η ε, απελευθέρωση των αγορών, σαν συνέπεια είχε, να βρεθούν άνεργοι χιλιάδες άνθρωποι. Η σουηδική βιομηχανία των μεταφορών δεν μπόρεσε να παραμείνει ανταγωνιστική σε σχέση με ξένες εταιρείες. Καταστροφή λοιπόν για την οικονομία μας και τις μεταφορές μας και μπορούμε πιστεύω να προβλέψουμε ότι μέσα σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν εθνικοί μεταφορείς, μεταφορικοί φορείς στην Σουηδία. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά σίγουρα μόνο την Σουηδία. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση. Και όσον αφορά το βάρος, αλλά και όσον αφορά το μήκος των βαρέων φορτίων, των φορτηγών ε, που κυκλοφορούν στους δρόμους μας, καθώς είναι όλο και πιο μεγάλα σε μήκο και όλο πιο βαριά τα φορτηγά αυτά. Είναι πολύ σημαντικό η κάθε χώρα να έχει το δικαίωμα να διατηρεί τους εθνικούς της κανόνες για να διαχειρίζεται αυτές τις οδικές μεταφορές που είναι όλο και πιο βαριές. Από την ιδιωτικοποίηση βλέπουμε όλο και πιο καταστροφικές συνέπειες γιατί θέλει κανείς όλο και περισσότερο κέρδος αλλά με όλο και λιγότερες επενδύσεις. Έχουμε στο παρελθόν ζήσει ένα αποτελεσματικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα δίκτυο όμως το οποίο από την ιδιωτικοποίηση και μετά δεν είναι καλό και δεν είναι δυνατόν πια να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Επικρατεί λοιπόν ένα χάος. Και αυτό είναι ο κανόνας περισσότερο παρά η εξαίρεση. Το ίδιο βλέπουμε να επεκτείνεται σε φαινόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εγώ την ιδιωτικοποίηση την είδα, την έζησα με τα δύο μου τα μάτια και δεν μπορώ να πω ότι είχε καλά αποτελέσματα στην Σουηδία και γι' αυτό δεν τη συνιστώ πουθενά στην Ευρώπη. Vielen Dank, Peter Lundgren. Und jetzt Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούντκβεν και τώρα πάλι ο Πρόεδρος. Μετά θα έχετε ακόμη ένα γύρο ερωτήσεων. Γι' αυτό θα χρειαστούμε αρκετό χρόνο, αλλά θέλουμε βέβαια και συγκεκριμένε ερωτήσει. Χωρί να είστε υπερβολικά δελεχεί, θέλουμε συγκεκριμένε απαντήσει σε ερωτήσει. Έχετε τον λόγο. Μάλιστα. Ευχαριστώ καταρχήν όλους τους συντονιστές που έθεσαν τις ερωτήσεις και στην Ιταλική Προεδρία. Καταρχήν να πω κάτι γενικό. για το τι καθοδηγεί και κινητοποιεί, παροτρύνει την Ιταλική Προεδρία για αυτό το εξάμεινο. Από πλευράς όλων σας ε, υπάρχει η συνείδηση η γνώση ότι δεν αρκούν πλέον τα προγράμματα, πρέπει να περάσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις να υλοποιηθούν τα προγράμματα τα οποία έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ επειδή βρισκόμαστε εδώ και μιλάμε ε, για το θέμα των συνδεδεμικών μεταφορών, την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, τα λιμάνια, ε, θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μα, των επιχειρήσεών μα, των οικογένειών μα. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένοι τρόποι εφαρμογής και υλοποίησης πλέον αυτών των προγραμμάτων τούτου λεχθέντος δηλαδή, ότι δηλαδή δέχομαι ε, ότι το αίτημα αυτό από πλευρά σας ότι η Ιταλική Προεδρία δηλαδή πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο συγκεκριμένα γιατί βρισκόμαστε επιπλέον στις αρχές της νέας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σημαντική αυτή η έξι μήνες διότι μπορούν να βοηθήσουν το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν να καθορίσουν τη ζωή των επόμενων πέντε ετών, να υπαγορεύσουν, να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές, να είναι ένα κίνητρο για να δούμε πώς η Ιταλική Προεδρία θα μπορέσει σε συγκεκριμένη, ε, με συγκεκριμένες πράξεις να μεταφράσει το αίτημα αυτό. Βεβαίως η τραγωδία της Ουκρανίας ε, ε, έπληξε τους πάντες, προσωπικά αλλά και ως κυβερνήσεις και θεσμούς. Βεβαίως όχι μόνο το, η δραματικότητα των όσων αλλά και το Εγγονώσω ότι θέτει τόσα ερωτήματα. Από μια πλευρά θέλουμε συγκεκριμένε να γνωρίζουμε όλη τη την, την πρόθεση να συσταθεί άμεσα μια διεθνή Επιτροπή έρευνα που θα διερευνήσει τα αίτια της κατάρρευσης του μαλαισιανού αεροσκάφους. Αυτό βεβαίως που εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι να θέσουμε αυτό το ερώτημα, να επαληθεύσουμε, και νομίζω αυτό ήταν και το, η ουσία της ερωτήσεώς σας, τη σχέση που έχει αυτή η τραγωδία με το πακέτο για τον ενιαίο ουρανό και ε, τη της ε, νομοθεσία ΕΜΣΑ. Η ασφάλεια των, ουρανών, των ευρωπαϊκών ουρανών είναι εγγυημένη. Η δυνατότητα συνεργασίας πρέπει να αυξηθεί στο ΛΕΝ και περισσότερο να υλοποιούνται κοινοί και ενωτικοί κανονισμοί. Αυτό ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Αυτό νομίζω είναι το θέμα που ακόμα μια φορά θα πρέπει να μας απασχολήσει, ακόμα και αν έμεσα μας φτάνει λόγω αυτής της τραγωδίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, τα άλλα ερωτήματα που έγιναν για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, για την, τον αργό ρυθμό της υλοποίησης του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ακριβώς αυτή την κατεύθυνση ε, ε, μας δείχνουν επίσης ότι δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε και να ξεπεράσουμε κυρίως στο Συμβούλιο τους διχασμούς που υπάρχουν ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και υλοποίηση όλος ιδιαίτερος όσον αφορά τα επίπεδα ασφάλειας ε, στις ε, αεροπορικές μεταφορές και να υπάρξει ε, επαρκή συντονισμός στην εναέρια κυκλοφορία. Να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν επιβραδύνει και ξέρετε σε τι αναφέρομαι, την ενεργοποίηση των FAB, δηλαδή των λειτουργικών τμήματων του εναέριου χώρου και έχουμε δηλαδή να διαπραγματευτούμε για το ΣΕΖΑΡ και για το ΕΑΖΑ, τους δύο κανονισμούς. Αυτά μας αναλογούν ως Προεδρία της Επιτροπής του Συμβουλίου με συγχωρείτε, Μεταφορών και αυτά μπορούμε άμεσα να τα κάνουμε. Προφανώς υπάρχουν φυσικά και όλα εκείνα που οφείλουμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πολιτική, ως κυβερνήσεις ε, ε, και όσον αφορά βέβαια αυτή την ε, τεράστια τραγωδία που συνέβη. Τώρα το κοινό θέμα γιατί επαναλήφθηκε αυτή η ερώτηση σε σχεδόν όλες τις παρεμβάσει και ακούστηκε και το τέταρτο συνδεδομικό πακέτο. Και εδώ, και πιστεύω δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε την τεράστια εργασία του Ευρωκοινοβουλίου στην τελευταία θητεία και τη δυσκολία να ε, προχωρήσουμε βήμα-βήμα συγκεκριμένα μπροστά ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Η ανησυχία σας είναι προφανώς το να γίνουν συγκεκριμένα βήματα ώστε να υλοποιηθεί αυτό το πακέτο. Η εργασία που έχει γίνει για το τεχνική, τεχνικό πυλώνα και από την Κομισιόν και από την ειδική ομάδα του, Ελλάδα, Ελλάδας, ε, της Ελληνικής Προεδρίας, ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί οδήγησε στον ορισμό των ε, τριών πυλώνων για το τέταρτο συνδρομικό πακέτο και επέτρεψε και στην Κομισιόν να έρθει, σε, να φτάσει μάλλον σε μια κοινή θέση για το τεχνικό πυλώνα. Στόχος της Ιταλίας φυσικά δεν είναι να τροχοπεδίσει οτιδήποτε, αντιθέτως να δώσει τη συμβολή της ώστε σε αυτό το, σε επιτυχή του τεχνικού πυλώνα να μπορέσουμε να φτάσουμε σε συγκεκριμένους ορισμούς, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και να μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε και σε πορίσματα. Η παρατήρηση που εμείς κάνουμε ως Προεδρία και πιστεύω πως ε, τη σημερινή συμμερίζεστε κι εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο, σε αυτή την Επιτροπή. Ε, ότι είναι ότι στο Συμβούλιο θα πρέπει, ενώ ορίζεται ο τεχνικός πυλώνας, δηλαδή μας δίνεται ένα συγκεκριμένο στόχος, ε, θα πρέπει να έχουμε το στένος, το θάρρος, ακόμα και για τα ε, ερωτήματα τα οποία θέσατε κάποιοι από εσά που παρενέβητε, να ξεκινήσουμε και να ορίσουμε το βασικό θέμα που είναι, το, ενός πακέτου, που είναι η διακυβέρνηση. Από τη στιγμή που έχουμε συνδέσει και έχουμε προσαρμόσει όλες μας τις υποδομές τεχνικές, ώστε η Ευρώπη να είναι ενωμένοι από τους ε, σιδηροδρομικούς διαδρόμους, πώς θα διακυβερνήσουμε την πρόσβαση, πώς θα ορίσουμε τα δημόσια συμφέροντα κάθε χώρας, πώς θα ρυθμίσουμε τον ανταγωνισμό, πώς θα ξεκινήσουμε να ορίσουμε ποιοι είναι οι κοινοί κανόνες, κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε αυτό. Αντιθέτως, είναι ακριβώς καθήκον της πολιτικής και των κυβερνήσεων, αν πιστεύουμε στην Ευρώπη και στο Κοινοβούλιο, να έχουμε το στένος να βρούμε τα κοινά σημεία, όχι τα σημεία που μας διχάζουν. Ή ο τεχνικός πυλώνας πρέπει να προχωρήσει και να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη συζήτηση στο Συμβούλιο και με το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά τον πολιτικό πυλώνα με αυτό το στόχο. Ε, προέκυψαν από τις δικές σας παρεμβάσεις οι ανησυχίες που υπάρχουν. Ότι δηλαδή το πρώτο αφορά ότι η απελευθέρωση μιας αγοράς δεν θα πρέπει να ε, ε, οδηγήσει στην εξάλληψη κάποιων δημοσίων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες και ουσιαστικές για ορισμένες χώρες και ορισμένες περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει το να μιλήσουμε για τον τεχνικό πυλώνα, να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Συγκεκριμένο στόχος της Προεδρίας μας είναι στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου να γίνει μια πρώτη πολιτική συζήτηση ανάμεσα σε όλα τα κρατημέλη, όπου θα προκύψουν, θα συζητηθούν όλες οι ανησυχίες, τα απαραίτητα στοιχεία που κάθε χώρα θα θελήσει να δώσει για τον ορισμό του πολιτικού πυλώνα. Με τρόπο ώστε στο τέλος του εξαμήνου να μπορέσουμε όχι να ολοκληρώσουμε το πολιτικό πυλώνα, γιατί θα, εμείς θα μπορέσουμε μόνο να ολοκληρώσουμε τον τεχνικό πυλώνα, αλλά να αρχίσουμε να έχουμε τις ε, συνιστώσεις ορισμένων βασικών θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση του τετάρτου σιδηροδρομικού πακέτου. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν λάθος από πλευρά της Ιταλικής Προεδρίας να μην προχωρήσει ενώ ολοκληρώνεται ο τεχνικός πυλώνας να μην προσπαθήσει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας λοιπόν, τεχνικός πυλώνας, έναρξη των διαπραγματεύσεων, έναρξη των συζητήσεων ανάμεσα στους υπουργούς για τη διακυβέρνηση, τον πολιτικό πυλώνα και την υπηρεσία τοπικής, τοπικών μεταφορών. Πολύ συγκεκριμένο και τεχνικό το πρόβλημα. Τώρα, συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά ας πούμε για τα δίκτυα TNT δεν υπάρχει πρόθεση, ίσως να μην εξηγήθηκα καλά. Δεν έχουμε πρόθεση να αλλάξουμε τους ορισμούς. Εδώ έχουμε κάνει μια πορεία από το 2008 Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα μπροστά. Ε, το πρώτο ήταν να οριστούν οι προτεραιότητες. 100 προτεραιότητες, όχι μία και δύο. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ ε, το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιό να μεγάλα βήματα μπροστά και το Συμβούλιο επίσης όσον αφορά τον ορισμό των ε, διαδρόμων και τα δίκτυα, για τα δίκτυα TNT γιατί έτσι ορίστηκαν οι προτεραιότητες. Τώρα, η μετάβαση που εμείς αναφέρουμε και μεταξύ άλλων ε, το λέω και για εκείνη την ερώτηση πώς αυτή η μεγάλη διάδρομη αυτά τα τεράστια έργα που είναι τόσο απαραίτητα και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων. Ποιος ήταν ο στόχος των δικτύων TEN-T. Από τη μια πλευρά η Ευρώπη να είναι όλα είναι και πιο ενωμένη. Από την άλλη να ανταπεξέλθουμε στην πρόκληση του, του, του σιδηροδρόμων, ποιότητα ε, περιβαλλοντική, ποιότητα της ζωής στην Ευρώπη, ανταγωνιστική πρόκληση του επιχειρηματικού μας συστήματος. Αυτήν θα, σε αυτήν θα ανταποκριθούμε μεταφέροντας τις μεταφορές από το γαουτσούκ στο σίδερο, από τους τροχούς στις ε, σιδηροτροχές. Έτσι Λοιπόν, εντοπίστηκαν οι προτεραιότητε, αλλά τώρα πρέπει να εντοπιστούν και οι κατάλληλοι πόροι, απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση όλων αυτών των προτεραιοτήτων και τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ε, θέλουμε λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά, γιατί είμαστε πεπισμένοι σήμερα ότι οι επενδύσει ε, που γίνονται για τις υποδομές δεν είναι κόστος, δεν είναι δαπάνη. Είναι μεγάλος πόρος για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Πρέπει όλοι να ε, δεσμευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και μια τελευταία παρατήρηση και κλείνω, Πρόεδρε, όσον αφορά την την θέρμανση του πλανήτη. Θυμίζω πως ακριβώς αυτή είναι η πρόκληση που όλοι μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είναι δυνατόν να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Ε, όπως είπε και ο πρόεδρος Ρέντς, είναι μια πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη να καταπολεμηθεί η, η θέρμανση του πλανήτη. Ε, Ακριβώς πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή και προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε με συγκεκριμένους πόρους, με αλλαγή συμπεριφορών, με τη δημιουργία υποδομών που θα ανταποκρίνονται σε, αυτές, σε αυτό το στόχο. Και δεν είναι τυχαίο που το άτυπο Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά, γιατί είναι ένα Συμβούλιο Μεταφορών και Υποδομών, ωστόσο θα αντιμετωπίσει σε διάλογο και με τους δημάρχους των Ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών πόλων θα ασχοληθεί και με το θέμα της κινητικότητας. Στα αστικά κέντρα. Γιατί εκεί έχουμε μεγάλη προκλήσει. Έχουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ούτω καθεξής. Μεγάλες προκλήσεις. Στα αστικά κέντρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλούς συναδέλφους που στον το λόγο. Δυστυχώς όμως πρέπει να τον περιορίσω, να περιορίσω το χρόνο σας σε ένα λεπτό και διαβάζω τα ονόματα. Herr de Grandes, Herr Bach, Herr Riquet, Herr Andersen, Frau Senalova, Herr Zelitska, Herr Koch, Frau Auto, Aito und Frau Darato. D'Amato und dann noch Boriba. Und dann ist die, weiß noch και, και ακόμη ένας συνάδελφος παρακαλώ. Και εγώ θέλω βέβαια να κάνω τις ερωτήσεις μου. Κλείνω τον κατάλογο. Αρχίζουμε με τον κύριο Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Λούπη, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε και σας ευχαριστώ και για αυτά που μας είπατε για την τραγωδία του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών που έλαβε χώρα στην Ουκρανία. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα στην πρώτη μας αυτή συνάντηση και στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο να εκφράσετε τη διαμαρτυρία σας για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα στην τραγωδία αυτή. στην αρχή ε, η τοποθεσία της τραγωδίας ήταν ξέφραγο αμπέλιο. Ο καθένας μπορούσε να μπαίνει, να βγαίνει, να εξαφανίζει αποδείξεις, ε, να απομακρύνει κάποια, κομμάτια από το αεροπλάνο ή οτιδήποτε άλλο στοιχεία. Θα πρέπει αυτά να τα επισημάνετε. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τις ενέργειε μεταφορές αλλά και τις εσωτερικές απλωτές οδούς, διαπιστώνουμε πολύ συχνά στους τομείς αυτούς κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεν θα πρέπει ο μοναδικός μας προσανατολισμός και η αιμονή μας ιδέα να είναι το κέρδος. Θα πρέπει να βελτιώσουμε και την οργάνωση, την επιμελητεία. Γιατί να μην λάβουμε υπόψη και το οικολογικό φορτηγό. Θα προχωρήσουν οι προσπάθειες στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Όταν εργαζόμουν στο χώρο των αερομεταφορών με είχε συγκλονίσει πριν από χρόνια μία σύγκρουση αεροπλάνων στον αέρα πάνω από τον ενέργειο χώρο της Ιουγκοσλαβίας. Ατύχημα ήταν, δεν ήταν ασκεμένη πράξη. Η συγγήτρια επίσης ήμουνα ως ε, βουλευτή στη συνέχεια για την ασφάλεια των αέριων μεταφορών μετά την 11η ε, Σεπτεμβρίου. Με συγκλονίζει λοιπόν το γεγονός ότι η τραγωδία της, ε, των μαλισιανών αερογραμμών οφείλεται σε σκεμμένη πράξη και όχι σε ατύχημα και ότι υπήρξαν κάποιοι που πάτησαν ένα κουμπί για να καταρρύψουν το αεροσκάφο. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον Υπουργό να ε, συζητήσει επανερχόμενο στο Συμβούλιο με τους ε, συναδέλφους του στις μεταφορές για να συζητήσουν και το θέμα της ειδωνοβλεπτικής συμπεριφοράς των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ε, σειραίουν, στέλνουν ε, τους απεσταλμένους τους στο χώρο της ε, τραγωδίας για να καταγράψουν στο δυνατόν πιο φρικιαστικές σκηνές. Επίση, πιστεύουμε κύριε Υπουργέ ότι θα, μπορέσουμε να θα ήταν καλό να προχωρήσουμε στου ενιαίου Ευρωπαϊκού ουρανού και το ΣΕΖΑΡ, αλλά βλέπουμε ότι πολιτική βούλη δεν υπάρχει. Έστω λοιπόν να εφαρμοστούν τα ισχύοντα και να καταπολεμήσουμε τα ιδιαίτερα συμφέροντα ορισμένων. Η Βρετανία υποστηρίζει τους ενιαίου Ευρωπαϊκού εθέρες, φαντάζομαι ότι και η Ιταλία. Το ίδιο γι' αυτό περιμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στη θητεία σα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, με ιδιαίτερη χαρά άκουσα την ομιλία σας και ε, πολύ συχνά ακούω τέτοιες εισαγωγικέ ομιλίες ε, από τις ε, Προεδρίες και διδάχθηκα δύο κοινά. Καταρχήν έχουμε το σταθερό τμήμα που επαναλαμβάνεται από τις διαδοχικές Προεδρίες αλλά δεν θα ε, γίνεται και πολλά γιατί έχουμε στο μεταξύ τις θερινέ διακοπέ και μετά τέσσερι μήνε πριν τι χριστουγεννιάτικε διακοπέ. Δεν θα έχουμε πολύ καιρό λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την τραγωδία, καταρχήν ε, ε, δεν ήταν τραγωδία, δεν ήταν απλώς αεροπορική τραγωδία, ήταν κατάρριψη αεροσκάφους. Θα πρέπει να μας πει ο Επιτροπός τι έκανε η υπηρεσία για την, οργανισμός για την ασφάλεια των αεροματοφορών, τι έκανε η Eurocontrol δεν έπεσε από μόνο του το αεροσκάφο. θα πρέπει να δοθούν κάποιε εξηγήσει. Δεν έχουμε ούτε ε, ένα εξάμεινο για να ελοπίσετε τι μακρόπνε προθέσει. προθέσεις. Επίσης, ε, το θέμα των ε, οδηγών των επαγγελματικών φορτηγών. Τι γίνεται με τις διανυκτερεύσει και όλε αυτές τι σχετικέ. Ε, ρυθμίσεις, επίσης διασυνοριακές μεταφορές. Ε, κάτι γίνεται στη Γαλλία, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις προσπάθειές μας, ώστε το επόμενο εξάμεινο να έχουμε απτές ε, προσπάθειες και αποτελέσματα, για να μπορούμε να πούμε Ιταλική Προεδρία και ο υπουργό Λούπη το Α και το Β συγκεκριμένο στοιχείο έκαναν κάτι επιτυχημένο και είχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ και εμείς αυτό ευχόμαστε βέβαια όλοι. Ο επόμενος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Μεταφορών και Υποδομών, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Ιταλό Υπουργό και να του ευχηθώ καλή επιτυχία για την Προεδρία και καλή τύχη για το επόμενο εξάμεινο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για, για την ανάλυση και την παρουσίαση που μας κάνατε των Ιταλικών προτεραιοτήτων φάνηκε ότι οι μεταφορές ε, βρίσκονται σε ένα κύριο σημείο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων, αλλά ταυτόχρονα οι μεταφορές ε, είναι σημαντικός τομέας για την ε, οικονομική ανάπτυξη αλλά και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Τα επισημάνατε όλα αυτά στην ομιλία σας οι μεταφορές θα πρέπει να έχουν σαφή προσανατολισμό. Η πολιτική των μεταφορών θα πρέπει να διέπεται από μια συγκεκριμένη στρατηγική προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ε, πρόσφορο επιχειρηματικό κλίμα που θα προσελκύει και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης ε, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν ε, στις διάφορες περιφέρειες και τα κράτη-μέλη και να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των περιφερειών. Εγώ κατάγομαι από νησί και η συνθήκη του Μάστριχτ έχει χαρακτηρίσει αυτή την περιοχή μαζί με άλλες ως εξόχως απόκεντρη περιοχή. Κατάγομαι από τη Μαδέρα, που είναι ένα νησί που παραλαμβάνω ανήκει στην κατηγορία των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Τέτοιες περιοχές έχουν Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία. Έχουν ιδιαιτερότητες λοιπόν αυτές οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και αυτές οι ιδιαιτερότητες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έχετε ένα λεπτό διακόπτει ο ε, ωραία, έρχομαι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ποια είναι η θέση της Ιταλικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά... Δυστυχώς... Όχι, λυπάμαι, πρέπει να σας διακόψω. Δεν μπορείτε να μιλήσετε περισσότερο. Έχετε εξατλήσει το χρόνο σας. Ο επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Για την οικονομική κατάσταση των Λιβανιών, συμπληρώνει η ομιλήτρια, ο κύριος Γκράντε Πασκουάλ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Λούπη. Η Ισπανική αντιπροσωπεία ε, του ΕΛΚ ε, ανεπιφύλακτα και αμέριστα συμμερίζετε τις προτεραιότητες σας. Θα ήθελα με τηλεγραφικό τρόπο να αναφέρω συγκεκριμένα σημεία. Καταρχήν είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση των διαφόρων διαδρόμων και αξώνων. Είναι πολύ σημαντική η ανάγκη πιο ελαστικής χρήσης των κρατικών και δημόσιων κονδυλίων για να χρηματοδοτήσουμε διασυνοριακά προγράμματα. Μας άρεσε ιδιαιτέρως η περιγραφή που κάνατε για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο που το χαρακτηρίσατε ολοκληρωμένο, ενιαίο. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο τεχνικό πυλώνα. Είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε και να συνεχίσουμε τις ε, ε, συνομιλίες και για το πολιτικό σκέλος του σιδηροδρομικού πακέτου. Λιμάνια, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, θα πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στην πολυτροπικότητα, στις μεταφορές με πολλαπλά μέσα. Θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές ε, οι λιμενικές υπηρεσίες και επίσης να εξασφαλιστεί μια διαφάνεια για να ενταχθούν και οι λιμενικές και οι θαλάσσιες μεταφορές, τις πολυτροπικές μεταφορές και φυσικά και οι συνδρομικές μεταφορές πολύ σημαντικές. Αμέριστη λοιπόν ανεπιφύλακτη υποστήριξη όχι μόνο στην Ιταλική μελωδία και τη μουσική αλλά και στο κείμενο, στο λιμπρέτο, σε αυτά που μας είπατε σήμερα για την Ιταλική Προεδρία. Ευχαριστώ και με χαρά ακούω τα όσα λέτε για την... Ε, περιμένω να ακούσω μάλλον για τον πολιτισμό και αυτά που μας φέρνει το Λουξεμβούργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, λέει ο κύριος Μπαχ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις ε, ε, εργασίες σας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα ενέργεια μεταφορές καταρχάς, με πολύ ε, κομψό τρόπο αποφύγατε να τοποθετηθείτε σε ορισμένα ζητήματα. Θα ήθελα να πω όμως ότι εμά μας ενδιαφέρουν όχι μόνο τα δικαιώματα των επιβατών αλλά και τα σλότ, οι χρονοθυρίδες και, όλες, ε, και όλη η προβληματική με την ε, ε, αντιπαράθεση με, γύρω από το Γιβραλτάρ και πώς νομίζετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μεταξύ των δύο κρατών. Στις ε, οδικές μεταφορές τώρα και την ασφάλεια. Έχουμε να κάνουμε προβλήματα τα οποία ακούστηκαν επί παραδείγματι ώρες ανάπαυσης και ύπνου των οδηγών, ε, επιβάρυνση στους δρόμους από τα gigaliners, τα πάρα πολύ μεγάλα φορτηγά. Ο Επίτροπος Κάλλας ε, πολύ συχνά παραπέμπει στα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν έχει έρθει νομίζω ακόμα η χρονική στιγμή ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις ενιαία στο θέμα αυτό και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από μια Ευρωπαϊκή Αποκεντρωμένη Υπηρεσία για τις Μεταφορές. Επίσης στους ε, σιδηροδρόμους, τα τεχνικά ζητήματα δεν μπορούν επιλειόμενα να επιτρέψουν την πρόοδο στο όλο πακέτο. κύριος Ρικέ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, προσπαθώ να είμαι και εγώ σύντομο. Καταρχά, ιδιαίτερα χαίρομαι για το γεγονό ότι υπογραμμίσατε και προβάλλατε τα προβλήματα των υποδομών τη ανάπτυξη ε, των προτεραιοτήτων που ορίσατε. Και ρωτώ το εξή. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με περιφέρεια περιφερειακή πολιτική, με προϋπολογισμό, με έρευνα, με πολιτική υποδομών και ενέργειας τηλεπικοινωνιών. Η Ιταλική Προεδρία σκέφτεται να συστήσει μια intergroup, μια μεικτή επιτροπή δηλαδή για να χειριστεί τα ζητήματα αυτά. Εγώ βλέπω ότι θα είναι δύσκολο μεμονωμένα κανείς να το λύσει, γιατί είναι πολύ κατακαιρματισμένα όλα αυτά τα θέματα. Και δεύτερη παρατήρηση για το σιδηροδρόμους. Από ό,τι βλέπω από τα όσα μας είπατε, το αντιμετωπίστε σε ένα όλον το θέμα των σιδηροδρόμων. Αλλά από την άλλη θα έπρεπε να είμαστε θέσει και να προχωρήσουμε στο βαθμό που μπορούμε στο κάθε θέμα χωριστά, αφαιρεπίν διακυβέρνηση κτλ. Και δεν θα έπρεπε να ξεκινήσετε τις επραγματεύσεις για τα τεχνικά στοιχεία που από ό,τι καταλαβαίνω μας λέτε ότι θα πράξετε. Ένα αναμονή πιο συγκεκριμένων ίσως ε, εξελίξεων ε, στα θέματα αυτά και ενδεχομένως και από πλευράς της βιομηχανία. Κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να ακούσω τι μπορεί να κάνει η Ιταλική Προεδρία για την ε, αντιμετώπιση των δυστυχημάτων των οδικών ε, υποτίθεται ότι πρόκειται να αντιμετωπιστούν ε, τα ποσοστά, οι στατιστικές των θανάτων από τροχέα, αλλά συγκεκριμένα μέτρα δεν βλέπουμε. Στο Ρωμένο Βασίλειο οπωσδήποτε δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα. Βλέπουμε μόνο περιορισμένη βελτίωση στα ε, στατιστικά στοιχεία των θανάτων από τροχέα. Ερωτώ λοιπόν την Ιταλική Προεδρία τι συγκεκριμένα έχει υπόψη. Η κυρία Σελάλοβα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ιταλικής Προεδρίας αλλά και για τις απαντήσεις που δώσατε στις προηγούμενες ερωτήσεις. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην τραγωδία των Μαλισιανών αερογραμμών και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Λιμπεράτσκι και να ρωτήσω και εγώ Πώς είναι δυνατόν ένα πολιτικό, πώς, τι γίνεται με ένα πολιτικό αεροσκάφος και γιατί επιτρέπεται η υπέρτισή του σε μια περιοχή που, ε, στην οποία λαμβάνει χώρα εμφύλιος πόλεμος. Τι έκανε η Eurocontrol. Επίσης, όπως είπε και η έχουμε μεγάλο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Πώς μειώσουμε αυτά τα τροχιά αντικείμενα. Και τι γίνεται με την ε, ίσπραξη, τη διασυνοριακή ίσπραξη των προστήμων, αλλά και το θέμα του e-call. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές και ελπίζω να ε, ολοκληρωθεί από την Ιταλική Προεδρία η ενσωμάτωση στο όχημα του e-call. Mm. Όντω ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, λέει κύριε Στέλισκα. Πολύ η ομιλία σα, φιλόδοξη και παρόλο που η βάση ε, για οποιαδήποτε αίσια έκβαση είναι μια σωστή τεκμηρωμένη ανάλυση, συμφωνώ με την ανάλυση σας, ήμουν όμως κάπως πιο απότομο και ομό. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε λειτουργική ε, εσωτερική αγορά μεταφορών, αλλά από τα στοιχεία που μας Αναλύσετε, διαπιστώνω ότι έχετε αντίληψη της κατάστασης. Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των μεταφορών και αντιμετώπιση των στενοπών ε, και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, πολύ σημαντικά θέματα και διαπιστώνω ότι ε, έχετε επίγνωση όλων αυτών των προβλημάτων. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι. Καταρχήν μακρόπνες φιλοδοξίες ε, και δεύτερον ενίσχυση και ουσιαστική υλοποίηση των υφισταμένων μέτρων και νομοθετικών διατάξεων. Γιατί υπάρχει κατακαιρματισμός, ε, υπερβολικός προστατευτισμός σε ορισμένες περιπτώσεις και πολλά προβλήματα. Φυσικά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να επομιστούν την ευθύνη, του, ευθύνη τους. Θέλουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ε, σωστή διακυβέρνηση και χρηστή οικονομική διαχείριση και διαφάνεια. Φυσικά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν ε, το βαθμό υλοποίησης των διαφορών διατάξεων. Θα πρέπει όμως ε, να αποσαφηνίσουμε στα κράτη-μέλη ότι αν υποβάλουν ε, σωστά σχέδια θα τύχουν και χρηματοδότηση, δεν μη θα χάσουν το δικαίωμά τους για χρηματοδότηση, αν δεν υποβάλουν τα κατάλληλα σχέδια. Επίσης, ε, θα πρέπει να διευκρινιστούν κάποιοι κανόνες για τις εταιρείε, αλλά για όλα αυτά θα έχουμε αρκετό χρόνο για διευκρίνηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έγινε στην πατρίδα μου ένα τροχαίο δυστύχημα το τελευταίο Σαββατοκύριακο με δέκα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ε, εμπλεκόμενα ήταν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό. Ένα λεωφορείο το οποίο δεν είχε ε, επαρκή συνθήκες ασφαλείας ως προς την πέδηση και του οποίου ο οδηγός δεν είχε ε, σεβαστεί τους κανόνες ανάπαυσης και ύπνου. Ίσως εάν, το εάν είχε σεβαστεί αυτούς τους κανόνες, να έχει αποφευθεί το τροχαίο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να επιβάλλουμε την εφαρμογή αυτών των κανόνων που ισχύουν εδώ και 10 τουλάχιστον χρόνια. Κυρία Αγιούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πλέον σαφέ. Ναι, εδώ βρίσκομαι. Μα το έχετε επαναλάβει ότι μία από τι κύριε προτεραιότητε του Ιταλικού εξαμήνου έχει να κάνει με την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών διαδρόμων. Πρόεδρε, ω πολίτη θα σα πω το εξή. Είναι πλέον προφανέ ότι δεν χρειάζονται αυτοί οι διάδρομοι. Υπάρχουν ένα σωρό μελέτες που το αποδεικνύουν, κυρίως ε, η σύνδεση λιον Υπάρχει η μελέτη του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, ας πούμε, που δείχνει ακριβώς ότι είναι άχρηστο ένα τέτοιο έργο και ότι θα ήταν προτιμότερο να γίνουν επενδύσεις σε, άλλες, ε, ε, σε άλλα σημεία όπου χρειάζονται έργο. Ενώ ο διάδρομος από την Ισπανία στην Ουγγαρία υπάρχει ήδη εκεί σιδηροδρομικό δίκτυο. Και σας αναφέρω την κοιλάδα του Τρεβίζο που ολοκληρώθηκε το 2000. Είναι πολύ σύγχρονος σιδηροδρομικός κόμβος, ωστόσο δεν οδήγησε στην ελάφρυνση του εισοδικής κυκλοφορίας. Ε, το αντίθετο μάλιστα. Να θυμίσω δε ότι με βάση μια πρόσφατη μελέτη στην Ιταλία το κόστος για την υψηλή ταχύτητα είναι 61 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις ε, τροχές μεγάλης ταχύτητας, δηλαδή ε, πολλαπλάσιο του κόστου σε άλλες ε, χώρες λόγω της διείσδυσης της μαφίας στις, στους διαγωνισμούς. Δεν θα ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για τα υπάρχοντα δίκτυα και να μην επιμείνουμε για την υλοποίηση μεγάλων έργων των οποίων η σκοπιμότητα αμφισβητείται και από ανεξάρτητους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Κυρία Αμάτο. Νταμάτο, διορθώνει η ίδια. Το τάραντο, το τάραντο συμπεριλήφθηκε στον θαλάσσιο διάδρομο με την Βαλέτα και με στους ε, χερσαίους διαδρόμους για τη σύνδεση Σκανδιναβικής με Μεσόγειο. Αυτό θα πρέπει να επιφέρει ωφέλη σε ολόκληρη την περιοχή. Υπάρχει όμως αμφιβολία, κυρίως η αμφιβολία για τον τουρισμό. Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Ιταλικού εξαμήνου έχουμε ε, και την διάδοση των καλών πρακτικών. Μέχρι στιγμής η περιοχή του αλλά και ολόκληρης της, ε, ε, ε, της, της περιοχής αυτής έχουν επιβεβαιωθεί από βιομηχανική ανάπτυξη χωρίς κανένα προγραμματισμό και πάλι θα τιμωρηθεί ο τουρισμός και ο πολιτισμός σε αυτή την πολύ σημαντική περιοχή. Μπορείτε να μας βεβαιώσετε ότι αυτό δεν θα συμβεί ακόμα μια φορά. Κύριος Κύριε Υπουργέ, λίγες σύντομες ερωτήσεις. Καταρχήν, είπατε ότι θέλετε να γίνει η ολοκλήρωση της, ε, και το άνοιγμα των ε, ε, μεταφορών επιβατών. Η Πολωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη για ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη τα επιχειρήματα της Πολωνίας κατά τη σύνταξη των νομοθετικών προτάσεων. Επίσης, το θέμα ε, της διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Είστε υπέρ του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, του unbundling, στον τομέα αυτό. Και τρίτη ερώτηση. Θα λάβετε υπόψη την δυνατότητα αποσύνδεσης διαχωρισμού κάποιων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Γιατί μερικές, μερικά τμήματα των διευρωπαϊκών δικτύων δεν έχουν καμία πιθανότητα να ολοκληρωθούν. Τέλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα, και δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ και θέλω να φερθώ σε τρία ζητήματα. Νομοθεσία καταρχάς θαλασσιών λιμένων για να ρωτήσω ποια είναι, ποιες είναι οι θέσεις ε, του Συμβουλίου ως προς την ιδιωτικοποίηση ορισμένων λιμενικών υπηρεσιών, επί παραδείγματι την πλοήγηση. Και ποια είναι η θέση ως προς τη σύγκρουση, τις, τριφές, τριβές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις ενισχύσεις προς τους λιμένες που οδήγησε τελικά στην αναβολή της πρώτης ανάγνωσης του θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. δεύτερο θέμα, η ατμοσφαιρική ρήπανση. Τι είδους προτεραιότητες θα δώσει η Ιταλική Προεδρία ως προς την φιλόδοξη, το φιλόδοξο στόχο της μείωσης της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης και πώς μπορεί να υλοποιήσει τουλάχιστον μέχρι το 2030 αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Κάλιτς. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα συνεχίσω, λέει ο κύριος τα στα κροατικά την ερώτησή μου. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, δώσατε μεγάλη έμφαση και σημασία στα προγράμματα υποδομών των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κροατία έχει απομονωθεί και έχει αποκλειστεί σχεδόν από τα δίκτυα αυτά ε, και έτσι δεν μπορούν να αποφεληθούν οι πολίτες της από τέτοια διευρωπαϊκά δίκτυα. Κροάτες που ζουν στον Ντούμπροβνικ και στην Έρετβα, στην επαρχία αυτή, είναι αποκομμένοι από την υπόλοιπη Κροατία. Επίσης θα πρέπει η πολιτική των μεταφορών να λάβει υπόψη και τις κλιματικές ελλαγές. Οι, οι πολίτες μερικές φορές θα πρέπει να θερύνονται να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Και για το σημείο αυτό θα, χρειαζόμαστε την βοήθεια και του Συμβουλίου και της Επιτροπής για να ολοκληρωθεί το φιλόδοξο σχέδιο της κατασκευής της, τράπεζ, της, τρα, της γέφυρας στη Χερσόνησο Πέλισσας που θα εξασφαλίσει τη σύνδεση και του Ντουμπρόβνικ με την υπόλοιπη Κροατία. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από μένα κύριε Υπουργέ. Θα σας ρωτήσω το εξή. Εάν είχατε την ανάκτικη 100 εκατομμύρια ευρώ και τη δυνατότητα μέσα σε δύο χρόνια να μειώσετε από 5 σε 2,5 ώρες την ε, οδική απόσταση από το Βερολίνο μέχρι τον Μπρέσλαο. Ή αλλιώς σε 10 χρόνια για 20.000 ευρώ να ανοίξετε ένα τούνελ από το, ε, μέσα από τις Άλπεις. Πού θα, πού θα ρίχναν το βάρος.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 Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ευρωβουλευτές που έθεσαν αυτές τις άριθμες ερωτήσεις, πολλές εκ των οποίων ε, θίγουν θέματα τα οποία ήδη ανέφερα στην εισήγησή μου αλλά και στις απαντήσεις μου στον πρώτο γύρο απαντήσεων. Ε, Φοβόμαι πως δεν θα έχω το χρόνο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα είναι χρήσιμες προτάσεις ε, θετικές για τη δράση μας διάρκεια του Προεδρείου, όπως θα είναι δίκαιο, νομίζω να είναι αυτός και ο στόχος της σημερινής ε, ακόρωασης. ανάμεσά μας και ανά, ανάμεσά μας την Προεδρία δηλαδή και το Ευρωκοινοβούλιο. Θα αναφέρω κάποια θέματα τα οποία τόσο στην έκθεση, στην εισήγησή μου όσο και στην πρώτη γύρω απαντήσεων δεν έθιξα. Το πρώτο θέμα το οποίο θα ήθελα όλος ιδιαίτερος να αναφέρω γιατί ήταν ένας από τους κεντρικούς ε, στόχους που είχαμε θέσει και ως Ιταλική κυβέρνηση αλλά θα πρέπει αυτό να αποτελέσει στόχο όλων των κυβερνήσεων στις Ευρώπη. Ε, και μάλιστα μία από τις πρώτες προτεραιότητες ήταν ο τεχνικός πυλώνας του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου που αφορά και την ασφάλεια, αφορά και τη συζήτηση που κάναμε στο πλαίσιο των Υπουργών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Όπως είπα λοιπόν, το νούμερο ένα είναι το θέμα της ασφάλειας ασφάλεια σε όλους τους τρόπους μεταφορών. Αεροπορικές μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, οδικές μεταφορές, αλλά και ε, μετακινήσεις γενικά. Ε, Τέθηκα σαν τα ερωτήματα για την ασφάλεια και για των οδικών μεταφορών, για τα θύματα των τροχιών ατυχημάτων, αλλά και την ασφάλεια των δημόσιων μεταφορών που μεταφέρουν ε, τον κόσμο στις διάφορες Περιοχέ τη Ευρώπη. Να θυμίσω ότι πέρσι στην Ιταλία υπήρξε, συνέβη μια τραγωδία πολύ σοβαρή, ίσως και πιο σοβαρή από τα όσα μας είπε ο κύριος Κόκο. 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ενό πολύ σοβαρού δυστυχήματος όπου ένα λεωφορείο που μετέφερε ανθρώπους που πήγαιναν σε μια εκδρομή τελικά το λεωφορείο δεν είχε σεβαστεί κανέναν από τους κανόνες ε, έλεγχος, κτέο, ασφάλεια κτλ. Το θέμα λοιπόν της πρόληψης, του ελέγχου και της ασφάλειας των δημοσίων μέσων μεταφοράς που κυκλοφορούν ε, στην Ευρώπη μεταφέροντας επιβάτες, το θέμα της ανανέωσης ε, του τροχαίου υλικού ε, γιατί έχουμε μέρη όπου ο μέσος όρος είναι 7 χρόνια ηλικία των μέσων ε, των οδικών μεταφορών, ενώ υπάρχουν ε, ε, χώρες όπως η Ιταλία όπου η ηλικία των μέσων οδικής μεταφοράς ανέρχεται στα 12-13 έτη. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην ασφάλεια αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, στη ρήπαση. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε προ αυτή την κατεύθυνση γιατί να είμαστε βέβαιοι ότι γίνονται οι έλεγχοι, να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει Ε, ότι μάλλον τα δημόσια μέσα μεταφοράς ε, θα εξοπλίζονται με τους ε, νέες καινοτομίες για το περιβάλλον αλλά και την ανανέωση των στόλων. Ε, πρέπει επίσης να φροντίσουμε για τη συντήρηση των δρόμων μας, γιατί 10% των ατυχημάτων οφείλεται στην κακή συντήρηση των ε, δρόμων. Ε, υπάρχει δέσμευση σε σχέση με τις επενδύσεις των μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την έκτακτη συντήρηση ή την προσαρμογή των υποδομών των δρόμων μας. Ακόμα και σε σχέση με τις πιο ευάλωτες κατηγορίες. Σκεφτείτε τους δρόμους στην Ευρώπη που έχουν κατασκευαστεί μόνο και μόνο με, τον τρόπο, με το παλιό τρόπο μεταφοράς, δηλαδή το αυτοκίνητο και δεν ε, προστατεύουν τους ε, ποδηλάτες και τους ε, μοτοσυκλετιστές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ανανεώνονται οι δρόμοι, να ανανεώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και αυτό είναι ένας από τους στόχους που έχουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί η πρόληψη γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Τέταρτο επίπεδο είναι η παιδεία και η ενημέρωση, η κατάρτιση, γιατί βέβαια πρέπει να δεσμευτεί ολόκληρη η Ευρώπη για την ασφάλεια, θα πρέπει να δοθεί δέσμευση από όλες τις χώρες για την παιδεία, την κατάρτιση, τη συμπεριφορά, γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Ωστόσο το θέμα της ασφάλειας για όλα μας τα μέσα μεταφοράς είναι το κύριο, είναι ο βασικός μας στόχος που πρέπει να θέσουμε και να έχουμε και τους απαραίτητους πόρους που θα τους αφιερώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε, και έτσι απαντώ, ε, δεν μπορούμε, έχουμε, έχουμε λίγο στους πόρους, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες, αλλά θα ήταν σφάλμα να αντιπαραθέσουμε τις επενδύσεις για τις την έκτατη συντήρηση για τη μικραία, μεσαία έργα και να ωφελήσουμε μόνο τα, τα μεγάλα έργα. Είναι απαραίτητα όλα αυτά, γιατί αυτά σε συνδυασμό μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες, εντάξει, και θα πρέπει να δώσουμε και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση, αλλά και ελέγχους που να κάνουμε για την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο θίγει και το οποίο επίσης είναι σημαντικό, ένας συνάδελφος ε, σας παρενέβη λέγοντας, μιλώντας μάλλον για το κοινωνικό ντάμπινγκ στον ε, τομέα της αεροπλοείας. Κοινωνικό ντάμπινγκ στον τομέα των μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για τις εναέρειες μεταφορές που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και για τις ε, οδικές μεταφορές. Κοινωνικό ντάμπινγκ στις μεταφορές τις οδικές όπου πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα. Γιατί έχουμε δύο μεταβλητές που διακυβεύονται εδώ. Η πρώτη αφορά τον αντίκτυπο που έχει το κοινωνικό ντάμπινγκ όσον αφορά την ασφάλεια. Σε όλους τις μεταφορές. Μείωση του κόστους σημαίνει μείωση των εγγύσεων όσον αφορά την ποιότητα και τις προδιαγραφές. Γι' αυτό μπορεί να είναι εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών. Ε, δεύτερο είναι ένα άλλο θέμα, όπου ότι δηλαδή εμείς ως Προεδρία, για το προεξάμεινό μας, αλλά πιστεύω πως είναι ο στόχος ολόκληρου του Ευρωκοινοβουλίου και όλων των κρατών μελών, να δώσουμε δουλειά στον κόσμο. Να δουλέψουμε για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Αλλά η απασχόληση θα πρέπει να προστατευτεί και να είναι μια απασχόληση αξιοπρεπή. Όχι μόνο ασφάλεια των θέσεων, αλλά και ε, αμοιβή. Κοινωνικό ντάμπινγκ λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και με θάρρος, με στένος. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να, σε, να κινηθούν σε διπλό μέτωπο. Έχουμε από τη μια ε, τις τεχνικές οδηγίες, τους τεχνικούς πυλώνες όλους τους τομείς. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την πτυχή ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, αλλά και από τις κυβερνήσεις που αφορά μια πτυχή που αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στοιχεία τα οποία δεν είναι αποκλειστικά τεχνικής φύσης, αλλά που εντοπίζουν και στόχο έχουν την ανάπτυξη και την κατεύθυνση, τη δρομολόγηση αυτών των προσπαθειών. Όσον αφορά και ολοκληρώνω το θέμα των λιμένων. Θα έλεγα ναι, ναι, ότι την επόμενη φορά θα... Εντάξει, πρέπει τώρα να τελειώσουμε, αλλά το θέμα των λιμανιών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είπα και στην εισήγησή μου, γιατί είναι ένα τομέα που ξέρουμε ότι από το λιμάνι μα περνάνε το 80% των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σημαντικό τομέα που πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χωρών αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτό το σύστημα και πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Στον κανονισμό, την οδηγία την οποία συζητάμε και θα έχουμε να τη συζητήσουμε και με το Ευρωκοινοβούλιο σίγουρα αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία του εξαμήνου αλλά και ολόκληρη τη θητεία πιστεύω. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, ευγενία σα, για τη διαθεσιμότητά σα, την υπομονή σα που με ακούσατε. Να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο για το χρόνο που μου ε, προσέφερε και θα απαντήσω και κατηδίαν για την επιλογή του φακέλου 1 ή του φακέλου 2 για το, το Ρήνο Λιών και τα υπόλοιπα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις. Στη δική μου δεν απαντήσατε την ερώτηση, περιμένω όμως να τα πούμε και κατηδίαν. Τρεις η ώρα λοιπόν με τον κύριο Κάλας για να καλωσορίσουμε και τους ε, νέους συναδέλφους και ευχαριστώ πολύ τους Ερμηνείς λέει ο Πρόεδρος που μας δώσατε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λούπη.